αυτή. Η μέρη διάταξη προβλέπει τώρα την έκθεση της κυρίας Ευαγγελίας Τζαμπάζη για την ψυχική υγεία. Παρακαλώ την εισηγήτρια, έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Συνειδητοποιούμε ότι προβλήματα ψυχικής υγείας βρίσκουμε συχνά και έχουν αντίκτυπο τόσο στην ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και κοινωνική ζωή των ατόμων και των οικογενειών τους, όσο και στην ίδια την κοινωνία με όρους ανθρώπινους και οικονομικούς. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Ένα στα τέσσερα άτομα θα αντιμετωπίσουν κάποια ψυχική διαταραχή η κατάθλιψη αποτελεί μία από τις πιο συχνές διαταραχές και έως το 2020 θα αποτελεί τη συχνότερη ασθένεια στον ανεπτυγμένο κόσμο. Στην Ένωση σημειώνονται κάθε χρόνο περίπου 59.000 αυτοκτονίες, 90% των οποίων οφείλονται σε ψυχικές διαταραχές. Ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες όπως παραδείγματος χάρη τα άτομα με αναπηρία έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουμε προβλήματα ψυχικής υγείας. σε μια ευρώπη επίσης η οποία γυράσκει η εμφάνιση νευροεκφυλιστικών διαταραχών γίνεται όλο ένα και συχνότερη. θα συμφωνήσουμε επομένως ότι η από αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζει η ψυχική υγεία είναι αναγκαία και μας αφορά όλους είναι υποχρέωση όλων να υπερασπιστούμε την ψυχική υγεία καθώς και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους αποτελεί ιδεολογική και πολιτική θέση σύμφωνα με την οποία το κράτος στηρίζει κοινωνικά και προστατεύει αυτούς που έχουν ανάγκη. Το πρώτο βήμα το αποτέλεσε η πράσινη βίβλος της Επιτροπής, το επόμενο βήμα έγινε με τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης μαζί για την ψυχική υγεία και την ευημερία, η οποία και καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ψυχική υγεία και την ευημερία. Σε αυτή την κατεύθυνση, η έκθεση για την ψυχική υγεία, η οποία υιοθετήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα, περιλαμβάνει μια σειρά από για την προώθηση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού, την καταπολέμηση του στίγματος, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού την ενίσχυση επίσης της προληπτικής δράσης και της αυτοβοήθειας και την παροχή υποστήριξης και επαρκούς θεραπείας στα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, τι οικογένειε και τους φροντιστές τους. Στην έκθεση τονίζουμε την ανάγκη για παροχή υψηλής ποιότητας προσιτών, προσβάσιμων, αποτελεσματικών και καθολικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και την ανάπτυξη σύγχρονης νομοθεσίας. Ζητούμε να δοθεί έμφαση στην κατάρτιση όλων των ατόμων στη θέση κλειδιά, ζητούμε τη διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση και δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, ζητούμε να δοθεί έμφαση στην πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας, μέσα από κοινωνικέ παρεμβάσεις ζητούμε από τα κράτη μέλη την ενδυνάμωση των οργανισμών που εκπροσωπούν τα ίδια τα άτομα με ψυχικά προβλήματα προτείνουμε τη θέσπιση μιας πλατφόρμας για την παρακολούθηση για την εφαρμογή του συμφώνου ζητάμε από την επιτροπή να παρουσιάσει τα συμπεράσματα των θεματικών διασκέψεων επισημαίνουμε την ανάγκη για ανάπτυξη κατάλληλων δικτών για καλύτερη εκτίμηση των αναγκών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. παράλληλα διατυπώνουμε προτάσεις στα πλαίσια των πέντε τομέων προτεραιότητας του συμφώνου. στο πλαίσιο αυτό τονίζουμε για την πρόληψη της κατάθλιψης και των αυτοκτονιών ότι απαιτείται η εφαρμογή πολυτομεακών προγραμμάτων καθώς και η ανάπτυξη δικτύων. Η ανάπτυξη ενός υγιού σχολικού κλίματος, η βελτίωση συνθήκων εργασίας, η ανάληψη μέτρων για τη βελτίωση ποιότητας ζωής και τέλος για την αντιμετώπιση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού τονίζουμε ότι απαιτούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Γι' αυτό, Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνέβαλαν με τις προτάσεις τους και να στείλουμε το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία είναι ύψιστο κοινωνικό αγαθό και οφείλουμε να εργαστούμε για την προαγωγή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, συγχαρητήρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην εισηγήτρια, την κυρία Τζαμπάζη, για την έκθεση αυτή ιδία πρωτοβουλία όσον αφορά την ψυχική υγεία. Πολύ σωστά η έκθεση υπογραμμίζει πόσο μεγάλη σημασία έχει η ψυχική υγεία και πόσο επηρεάζει την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός λοιπόν ότι δύο χρόνια μόνο μετά από ένα ψήφισμα που ήταν απάντηση στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίνει λοιπόν μια έκθεση δύο χρόνια μετά, δείχνει τη σημασία που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το θέμα. Και αυτό με κάνει εμένα να είμαι πιο αισιόδοξο. Σημαίνει ότι είναι γνωστή η σημασία που έχει η ψυχική υγεία για όλους τους τομείς υπήρξε υψηλού επίπεδου διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψυχική υγεία και τις επιπτώσεις της, κάτι το οποίο ανέφερε και η συγγήτρια. Και έτσι πιστεύουμε ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Εξάλλου πολλές χώρες μέλη έχουν φροντίσει να συμπεριλάβουν στρατηγικές ψυχικής υγείας ή προγράμματα δράσης, όπως για παράδειγμα στη Φιλανδία και στην Ουγγαρία. Επίσης, έχει συμπεριληφθεί το θέμα πολλές φορές ε, στη, στα σχολικά προγράμματα εκπαίδευσης. Οι εργοδότες επίσης όλο και περισσότερο γνωρίζουν τη σχέση που έχει η ψυχική υγεία με την παραγωγικότητα. Και είναι πολύ βασικό όντως να νιώθει κανείς καλά στη δουλειά του. Βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, Πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Δεν πρέπει να υπάρχει κίνδυνος για την ψυχική υγεία εξαιτία της ε, οικονομικής κρίσης. Τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να μπουν στον πειρασμό να μειώσουν τις δαπάνες τους για την ψυχική υγεία ή για τα συστήματα υγείας τους. επανερχόμενα στο παλιό τύπο άσυλα. Όμως, ιδιαίτερα για τους νέους, η ψυχική υγεία έχει τεράστια σημασία. Υπάρχει αστάθεια, υπάρχει ανησυχία, ανεργία και όλα αυτά αποτελούν μεγάλη απειλή για την ψυχική υγεία. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οργανώσει διάφορες θεματικές διασκέψεις για τις πέντε προτεραιότητες όσον αφορά την ψυχική υγεία. Οργανωμένα από κοινού με τις Προεδρίες του Συμβουλίου και τα κράτη-μέλη. Διάσκεψη για την ψυχιατρική φροντίδα θα οργανωθεί 29 Μαΐου από την Τσεχική Προεδρία. Η πρώτη θεματική θα είναι για την νεότητα στη Στοκόλμη. 29 και 30 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με τη Σουηδική Προεδρία. Δεύτερη θεματική διάσκεψη για την πρόληψη της κατάθλιψης και της αυτοκτονίας από κοινού με την Ουγγαρία το Δεκέμβριο. Πρώτο εξάμεινο 2010, η Ισπανική Προεδρία θα φιλοξενήσει θεματική διάσκεψη για την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων. Στη συνέχεια, είμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη όσον αφορά άλλες διασκέψεις για την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας, το στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει πολλές συγκεκριμένες προτάσεις που βοηθούν πολύ για την εξέλιξη και τις μελλοντικέ συζητήσεις που θα κάνουμε για το θέμα. Γιατί η έκθεση δεν λέει μόνο πόσο σημαντική είναι η ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποδεικνύει επίσης ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να δράσουμε στον τομέα της ψυχικής υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από τις προτάσεις στην έκθεση είναι να υπάρξει μία δομή για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Ψυχική Υγεία. Συμφωνώ ότι θα είναι θέμενη αξία εφόσον θα αξιολογούμε κάθε τόσο την πρόοδο που έχει γίνει σε σχέση με το σύμφωνο αυτό. Έτσι θα φροντίσουν να δούμε πώς στην πράξη μπορεί να μπει σε εφαρμογή μια τέτοια ιδέα. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την εισηγήτριά του για την τόσο καλή αυτή έκθεση ε, και τις τόσο σημαντικές συστάσεις που περιλαμβάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 10.30. Θα διαπιστώσατε ότι χαμηλώσαμε το φωτισμό της αίθουσας. Φαντάζομαι είναι για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Τέλεια, γιατί ε, τώρα στην ε, ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση Αντρέας Γιούρκ για τη συνέχεια που δόθηκε στα εθνικά σχέδια για την ενεργειακή απόδοση. Μια πρώτη